το νέο μέλος της Επιτροπής μας. Καλή επιτυχία, καλή δουλειά εδώ στην Επιτροπή μας. Πάμε τώρα στο σημείο παραδείγμα 7. Το κοινό έργο, ΙΜΚΟ και ΙΤΑ, σχετικά με την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών. Έχουμε μαζί μας την ε, πρόεδρο της ε, ΙΜΚΟ, γίνεται ε, με βάση τον φαινονισμό 55 Κάθε συνάντηση θα έχει διαφορετική ε, ημερήσια διάνταξη ε, και θα έχουμε μία τελική έκθεση ε, και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην συμπροεδρεύουσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάνκ για τον λόγο. Θα ήθελα λοιπόν να ανακοινώσω την έναρξη της συνεδρίασης. προβλέπεται μία ώρα ε, για, ε, να, ε, για το σχέδιο έκθεσης αυτό και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχόλια τότε η συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη θα εγκριθεί. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι η συγκεκριμένη συνάντηση μεταδίδεται μέσω του ίντερνετ, είναι e-meeting επίσης οπότε όλα τα έγγραφα θα τα βρείτε στο ίντερνετ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο πίσω στον συμπροεδρεύοντά μου. Υιοθετήθηκε λοιπόν η ημερήσια διάταξη, ε, μπορούμε να ξεκινήσουμε και θα ήθελα να δώσω αρχικά το ε, λόγο στους δύο εισηγητές, αρχικά στην κυρία Μόσκα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μια γενική εικόνα σχετικά με το λόγο, για ποιο λόγο μιλάμε ε, για τον συγκεκριμένο ε, κανονισμό. Υπολογίζεται στα 56 δισεκατομμύρια πωλήσει για το 2016 σε πολιτιστικά αγαθά και υπολογίζεται ότι γύρω στο 19% των πωλήσεων είναι, από, είναι παράνομα. Για αυτόν τον ε, λόγο, λοιπόν, ε, θέλουμε ένα πιο μόνιμο πλαίσιο ε, από το να επικεντρωθούμε σε μεμονωμένα περιστατικά, όπως συμβαίνει με τη Συρία και το Ιράκ. Ε, όσον αφορά αυτή την ε, πρόταση, η συζήτηση ήταν ε, πολύ έντονη. Λάβαμε γύρω στις 270 τροπολογίες και είναι ξεκάθαρο ότι οι περισσότερες πολιτικές ομάδες είναι υπέρ αυτής της πρωτοβουλίας. Είναι καιρός λοιπόν να ενώσουμε τις διάφορες θέσεις και να υπάρξουν συμβιβασμοί για την έγκριση αυτής της πρότασης. Από γενική σκοπιά η ομάδα μου υπερασπίζεται, υποστηρίζει την ε, συγκεκριμένη πρόταση για την αντιμετώπιση την παρα, της παράνομης ε, ε, πολιτιστικών αγαθών. Πρόκειται για μια επιχείρηση δισεκατομμυρίων που βλάπτει τους φορολογούμενους, χρηματοδοτεί επίσης τις εγκληματικές δραστηριότητες και την τρομοκρατία και στόχος μας θα είναι λοιπόν να υπάρξει η ορθή ισορροπία μεταξύ της υπεράσπισης της πολιτισμικής κληρονομιάς ε, και την ανταγωνιστικότητα της ε, αγοράς. Προτείνουμε λοιπόν συγκεκριμένα μέτρα ε, και, και παροχή βοήθεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ε, απαρτίζουν το 75% της αγοράς. Επίσης, χρειαζόμαστε μία ε, παράγραφο για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, με ένα ειδικό πλαίσιο για αυτές και να περιλάβουμε ένα κεφάλαιο για την επίδραση που θα έχει στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάτι το οποίο υποχρεούται να παρουσιάσει ο, ο Επίτροπος στο Κοινοβούλιο. Ναι, θα ήθελα επίσης να αναφέρω άλλα δύο ζητήματα όπως αφορά ε, το κοινό ηλεκτρονικό σύστημα όσον αφορά τη χορήγηση αδειών και να μειώσουμε τον ε, χρόνο ε, που απαιτεί, απαιτείται ούτως ώστε να ενημερώσει η Κομισιόν το Κοινοβούλιο. Ως συνεισηγητές δεν βρήκαμε συμφωνία όσον αφορά συγκεκριμένα τεχνικά ζητήματα. Θα Αθήνα να γίνει τροπολογία του παραρτήματος σχετικά με τον κανονισμό εξαγωγών ε, εάν ε, ε, επικεντρωθούμε σε μια εκτελεστική πράξη τότε απομακρυνόμαστε από την εμπειρία. Θα πρέπει όσον αφορά τα πιο πολύτιμα αγαθά το πλαίσιο των 100 χρόνων το οποίο συμβαδίζει περισσότερο με την UNESCO καθώς επίσης και ε, την ε, ενημέρωση των ε, των ε, διασαφιστών που έχουν μεγαλύτερη κοιότητα πάνω σε αυτό. Ε, η πρόταση δεν είναι ιδεολογική, ε, δεν θα μεταφέρει το εύρος στα πιο πολύτιμα αγαθά και θα διασφαλίσει το ίδιο επίπεδο προστασίας σε αγαθά, πολιτισμικά αγαθά τα οποία παράχθηκαν νωρίτερα από 250 χρόνια. Θα δώσουμε με αυτόν τον τρόπο ένα ακόμα εργαλείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του παράνομου εμπορίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τώρα ο συνεισηγητής ε, για την Ίνκο, κ. Ντάλτον. Ευχαριστώ πολύ. Θα υποστηρίξω τα όσα είπε η κυρία Μόσκα για την ε, συνεργασία μας. Τρία είναι τα βασικά σημεία αυτού του σχεδίου έκθεσης κατά την άποψή μου μάλλον, συγγνώμη, τα τρία βασικά σημεία είναι η χρήση του ψηφιακού κόσμου, ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οι διεθνεί προσπάθειε. Ε, οπότε θέλω να τα εντάξουμε όλα αυτά σε ένα πολιτικό πλαίσιο για την ψηφιακή προσέγγιση. Εμεί συμφωνούμε με την κυρία Μόσκα για μια ψηφιακή προσέγγιση των τελωνιακών διαδικασιών, ειδικότερα για τα πολιτιστικά αγαθά τα οποία μεταφέρονται για αισθητικούς λόγους, δεν παράγονται από κάποιον, απλά τα απολαμβάνουν οι κατοχοί τους. Οπότε χρειαζόμαστε την ψηφιακή αξιοποίηση ώστε να βοηθάει και τη δουλειά των τελωνίων. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ένα σημαντικό κομμάτι της αγοράς εργών αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πολύ μικρές επιχειρήσεις, πολύ ειδικευμένες εταιρείε ε, εμπορίου εργών Δεν είναι χώρος μεγάλων πολυεθνικών, είναι οικογενειακής επιχειρήσεις στην καρδιά αυτού του εμπορίου. Χαιρόμαστε λοιπόν που έχουμε κοινή προσέγγιση και για αυτό το σημείο βάσει της εμπειρίας ε, που έχουμε ε, και από την υποστήριξη προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουμε και σε εκθέσεις σας. Τώρα για την ανάπτυξη ικανοτήτων και την κατάρτιση προτείνουμε κάποιες βελτιώσεις στο κείμενο. Είναι σαφές ε, ότι η περιστολή της ροής μέσω προσπάθειών δεν θα επιλύσει το πρόβλημα, διότι δεν επιλύεται η πηγή του προβλήματος. Αυτό το αναγνωρίζουμε και οι δύο μας. Υπάρχουν πολλά προγράμματα με πολλά μουσεία της Ευρώπης ώστε να υποστηρίξουμε την προστασία των έργων τέχνης στις περιοχές σειράξεων. Με την περιστολή λοιπόν των εισαγωγών ε, ουσιαστικά ε, μόνο, αντιμετωπίσουμε μόνο ένα κομμάτι αυτού του παγκόσμιου προβλήματος δεδομένης της εξαιρετικής μας συνεργασίας ε, μέχρι στιγμής και τη συνεργασία μεταξύ των σιωδών. Πιστεύω ότι θα έχουμε προοδεύσει σε αυτή την πρόοδο την έκθεση πριν το καλοκαίρι. Οπότε, αλλά απομένουν κάποια δύσκολα ερωτήματα. Μια από τις βασικότερες δυσκολίες είναι το αντικείμενο. Τι χρειάζεται για να, προλάβουμε, για να αποτρέψουμε την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με τέτοιου τρόπους και ποια μέτρα θα ήταν αποτελεσματικά για το σύνολο του παράνομου εμπορίου. Το σχέδιο ε, πρόταση ε, αναγνωρίζει ότι αυτά τα δύο προβλήματα είναι διαφορετικά και απαιτούν διαφορετικέ λύσει. Εμεί πρέπει να το διατηρήσουμε αυτό το διτό χαρακτήρα, ότι η χρηματοδότηση τη τρομοκρατία χρειάζεται συγκεκριμένη στοχευμένη παρέμβαση ε, και διαφορετική από την αντιμετώπιση που έχουμε για το παρανομό εμπόριο. Θέλουμε λοιπόν να μην συμπεριλάβουμε στοιχεία τα οποία δεν αφορούν αυτή τη χρηματοδότηση τρομοκρατίας. Δεν θέλουμε να κάνουμε ρυθμίσεις βάσει μιας ρομαντικής άποψης ή κινηματογραφικής άποψης για το τι είναι το παράνομο εμπόριο. Δεν ξέρουμε πόσα ε, αντικείμενα, πόσα στοιχεία θα επηρεαστούν από αυτό γιατί οι εκτιμήσεις και από την Επιτροπή ή με άλλους παράγοντες ε, το πόσες άδειε θα χρειαστούν ε, κυμαίνονται από δεκάδες μέχρι χιλιάδες. Εμείς γνωρίζουμε από τις αναλύσεις των εξαγωγικών αδειοδοτήσεων που δίνονται υπό συγκρίσιμες συνθήκες ότι από 10 έως και 20.000 άδειε δίνονται ετησίως. Μιλάμε για χιλιάδες ε, αντικείμενα τα οποία πρέπει να εκτιμηθούν. Επίσης είναι σημαντικό να εξετάζουμε τις αιτήσει και όχι μόνο τις άδειες που έχουν χορηγηθεί, γιατί και οι αιτήσει, ακόμη και όταν έχουν απορριφθεί, χρειάζονται εκτίμηση. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση σε συγκεκριμένα κατόφλια και δείκτες, ώστε να ζητάσουμε καλύτερα τους πόρους μας και τις προσπάθειές μας. Να έχουμε μια λίστα επικίνδυνων χωρών μαζί με διάφορες προτάσεις ε, για τα ε, ορυκτά από σειράξεων και άλλα πλαίσια που έχουμε και σε άλλα νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως κανόνες για τις εξαγωγές πολιτιστικών αγαθών από τις ευρωπαϊκές χώρες. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να στοχεύσουμε τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αλλά να αποφύγουμε τις παγίδες ε, που θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι τελωνιακές αρχές για τις εισαγωγές κανονικών νόμιμων αγαθών και επίσης να συμπεριλάβουμε τις περιπτώσεις όπου απαιτούνται αποδεκτικά στοιχεία αλλά είναι δύσκολο να δοθούν. Ε, υπάρχουν κάποια αντικείμενα ε, τα οποία ανήκουν σε οικογένειες ε, για γενιές, μπορεί τα, κάποια πολιτιστικά ιδρύματα να μπορούν να αναγνωρίσουν ακριβώ την καταγωγή. Οπότε χρειαζόμαστε ένα πιο περιορισμένο φάσμα ώστε να δράσουμε πιο αναλογικά. Ε, κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρίς να πιαστούν όλοι σε ένα ε, δίκαιο, αδιάκριτο δίκτυ. Ένας άλλος τομέας που είναι σημαντικός είναι οι, αρχε... οι εξουσίες που δίνουμε στις αρχές ε, έχουν ήδη κάποιες εξουσίες, αλλά πρέπει να τους δώσουμε εξουσίες που να μην παραμείνουν στα χαρτιά ή σε ηλεκτρονικά αρχεία. η νόμιμη εξαγωγή ε, μπορεί να μην ε, τεκμηριώνεται με μια κλασική διασάφηση. Οπότε θα πρέπει να έχουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία της εξαγωγής. Εμείς θέλουμε λοιπόν η διασάφηση για τα πολιτιστικά αγαθά να επεκταθεί ώστε να υπάρχουν πιο συγκεκριμένα στοιχεία που να χρησιμεύουν στις τελωνίκες αρχές. Ε, ελπίζω αυτό να δώσει μια καλή εικόνα των δικών μου απόψεων για την πρόταση και αναμένω τα σχολεία σας. Thank you very much. And then I would like to give the floor. Σε ευχαριστώ πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στους και συζητητές και πρώτος ε, Ελκα Ιμκο Φερχάγιν Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, αρχικά στους, ε, όσον αφορά τους συνηγητές, θεωρώ ότι πρέπει να εργαστούμε ακόμα πάνω στην συγκεκριμένη έκθεση. Είμαι πολύ θετικά στα όσα ανέφερε ο κύριος Ντάλτον. Χρειαζόμαστε μία, ε, ήδη, ε, έχουμε ήδη μια μεγάλη προστασία όσον αφορά τα πολιτιστικά αγαθά τα οποία έχουν ε, έρθει παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χρησιμοποιούνται ως χρηματοδότηση τρομοκρατίας. Από την άλλη δεν θέλουμε να καταστρέψουμε την αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση πνίγοντας την, με την γραφειοκρατία Έχουμε ε, παραδείγματα ε, τέτοια. Θα υπάρξουν λοιπόν ε, σοβαρές δυσκολίες για τους μικρότερους εμπόρους και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και γι' αυτό το λόγο χρειάζονται ξεκάθαρες τροπολογίες σχετικά με το για ποιους ισχύουν όλα αυτά. Είναι σημαντικό να διαφοροποιήσουμε λοιπόν όταν μια χώρα έχει που είναι χώρα προέλευσης πολιτιστικού αγαθού έχει ένα αρκετά καλό καθεστώς προστασίας τότε μπορούμε πολύ εύκολα ε, να συνεργαστούμε με αυτό σε αντίθεση ε, με την περίπτωση ενός πολιτισμικού αγαθού όπου η προστασία πολιτισμικών αγαθών ε, δεν είναι τόσο καλή και ιδιαίτερω όταν αυτή η χώρα βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με αποτέλεσμα τα πολιτιστικά αγαθά να μην χαίρουν τη αναγκαία προστασία. Και εδώ νομίζω λοιπόν ότι ε, θα πρέπει να έχουμε μια ισχυρή προστασία ε, των πολιτιστικών αγαθών από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εισαγωγή τους ε, και γι' αυτό το λόγο θα θεωρώ ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν να δημιουργηθεί μια λίστα με χώρε σε εμπόλεμη κατάσταση για να λαμβάνεται υπόψη και να έχουμε από τη μία ε, την, ε, το πολιτιστικό αγαθό και την αγορά και από την άλλη την προστασία του πολιτιστικού αγαθού. Ευχαριστώ πολύ ε, και τον κύριο Βαλές από το EPP. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. υπάρχουν πολλά παραθυράκια σε αυτήν την πρόταση που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πρώτον, θέλω να επαναλάβω ότι ο ορισμός ε, περιλαμβάνει όλες τις ε, κατηγορίες ε, και τον περιορισμό των 250 χρόνων που έχει οριστεί για όλες τις ομάδες πολιτιστικών αγωθών. Δεν θεωρώ ότι αυτό το όριο είναι επαρκές. Είναι, είναι ο έλεγχος ε, μονάχα των πολιτιστικών αγωθών άνω των 250 ε, χρόνων θα έχει ως αποτέλεσμα έργα τέχνης ε, και μοναδικά τεχνουργήματα τα οποία έχουν κλαπεί θα μπορούν εύκολα να εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, όσον αφορά τις προτινόμενες κατηγορίες βλέπω κάποια προβλήματα. Ε, όπως για παράδειγμα, τι ορίζεται ως σπάνια συλλογή και ποιο θα είναι το όριο υλικό ηλικία όσον αφορά την απόκτηση αυτής της ε, ε, συλλογής. Ε, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι, ότι εξελίσσεται η αρχαιολογία και η ιστορία και κάτι το οποίο στο παρελθόν δεν θεωρούνταν πολύτιμο, τώρα ίσως να είναι κάτι το οποίο επιθυμούν πάρα πολλοί συλλέκτες. Έτσι λοιπόν το όριο για την κατηγοριοποίηση ε, των πολιτιστικών αγωθών θα πρέπει να είναι ευμετάβλητο. Ε, το άλλο θέμα αφορά την ε, χώρα πηγή σύμφωνα με το άρθρο 2. Πρόκειται για τη χώρα όπου δημιουργήθηκε ή ανακαλύφθηκε το αγαθό. Αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να αλλάξει και γι' αυτό το λόγο θα καταθέσω τροπολογίες. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι είμαι υπέρ ε, του ε, να εισάγουμε μια εισαγωγή ε, παράνομων εξαχθέντων πολιτιστικών αγαθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να υπάρχει και αυτή η λίστα για να προστατεύσουμε τις χώρες, τις χώρες από την χρηματοδότηση τρομοκρατίας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να προσεγγίσουμε αυτό το στόχο, θα πρέπει όμως να βρούμε ένα κοινό σημείο. Και τώρα από τους ληστές για την ΙΜΚΟ, ο κύριος Κον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές ε, για ε, την πρότασή τους ιδιαίτερως όσον αφορά τα παραρτήματα και εκεί περιλαμβάνονται διάφορα ε, θέματα. Θα πρέπει να ξέρουμε για ποια πολιτιστικά αγαθά μιλάμε ακριβώς, ε, ποιος, ε, τι ακριβώς θα ελέγχει ο διασαφιστής κατά την εισαγωγή τους, Κατά τη γνώμη μου λοιπόν ε, σε αυτό ε, το πλαίσιο δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε εκ νέου τον ε, τροχό. Υπάρχουν οι κατευθυντήριες της UNESCO, υπάρχουν τα ηλικιακά όρια, υπάρχουν τα ζητήματα τα οποία πρέπει να ελέγχονται και δεν θα πρέπει να απλοποιήσουμε μονάχα το το έργο των τελωνίων αλλά ταυτόχρονα και τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, κάτι το οποίο θα διευκόλυνε ε, περισσότερο. Ε, και προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται οι τροπολογίες που θα καταθέσω. Ευχαριστώ πολύ και εφόσον ο κύριος Κάμπελ δεν είναι εδώ, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Σελίμοβιτς από το Άλντε για την ΙΜΚΟ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι αρκετά δύσκολο όπως φαίνεται το θέμα αυτό, τόσες πολλές διαφορετικές απόψεις. Εγώ θα προσπαθήσω να σας δώσω τη φιλελεύθερη πλευρά. Είναι προφανές ότι το παράνομο εμπόριο αρχαιοτήτων εκτιμάται σε περίπου 6 δισεκατομμύρια ε, αμερικανικά δολάρια ετησίως. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Κοινοβούλιο και πολλά από αυτά τα χρήματα όπως αναφέρει και αναφέρεται υποστηρίζουν πράγματι και χρηματοδοτούν την τρομοκρατία. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε. Έχουμε ήδη ανταποκριθεί με κάποια έγγραφα σημαντικά, έχουμε ήδη μέτρα. Έχουμε επίσης ε, και νομοθεσία που ρυθμίζει τις εξαγωγές των πολιτιστικών αγαθών, αλλά υπάρχει ένα κενό ακάλυπτο, απουσία κανονισμού που να αφορά την εισαγωγή των πολιτιστικών αγαθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό τον λόγο καλωσορίζουμε τις προτάσεις της Κομισιόν. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε και τους ε, δύο εισηγητές ε, για το σχέδιο αυτό. Παρ' όλα αυτά το άρθρο 4 και 5 που είναι ο πυρήνας της πρότασης φαίνεται να μην μας βρίσκει σύμφωνος. Ο ένας από αυτούς θα ήθελε να δίνεται άδεια εισαγωγή σε όλα τα προϊόντα εισαγωγής ανεξαρτήτως του είδους τους. Ο άλλος εισηγητής θα ήθελε να στοχεύσουμε σε συγκεκριμένες απειλές, συγκεκριμένες χώρες. Εκεί συμφωνούμε με τον κύριο Ντάλτον. Η διασάφηση εισαγωγής πρέπει να είναι ομαλή, εύκολη στοχευμένη διαδικασία, να μην υπερφορτώνει τους εισαγωγείς ε, πολιτιστικών αγαθών, ειδικότερα όταν τέτοια αγαθά είναι απίθανο να χρηματοδοτούν την τρομοκρατία, που αυτό συμβαίνει στην πλειοψηφία του ουσιαστικά επίσης, θα πρέπει να δοθεί μέγιστη ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την απόψή μας ώστε να γίνεται διάκριση των αγαθών ε, ε, και σε ποια διαδικασία θα υποβάλλονται. Μου φαίνεται ότι έχουμε εδώ μια προσέγγιση γενική για όλα στις περιπτώσεις ε, κάτι κατάλληλο για αυτή την περίπτωση, ειδικότερα αν σκεφτεί κανείς τους διάφορους τύπους αγαθών, τους διάφορες οδούς μεταφοράς, ε, ε, τους οικονομικούς φορείς και τη διαφοροποίησή τους. Άλλοι είναι πιο επικίνδυνοι από άλλους, οπότε τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα, αφού η τελωνικοί έλεγχοι γίνονται σε εθνικό επίπεδο. Πέραν αυτού, ε, θα υποβάλλουμε κάποιες τροπολογίες πολύ καλές ε, για αυτά τα σημεία. Οι διαδικασίες στο άρθρο 4 και 5 πρέπει να είναι ηλεκτρονικές, να χρησιμοποιούνται εύκολα και να υπάρχουν πριν τεθεί σε ισχύ η Επιτροπή. Η Επιτροπή δεν λέει τίποτα για το πώς η διαδικασία θα έχει στην πρακτική και δεν φανταζομαι ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα χρειαστεί να ξαναδιαβάσουν να διαβάζουν χαρτιά για να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία. Επίσης, ε, αρρωγή προς τις τρίτες χώρες για να τις ενημερώσουμε για τους κινδύνους και τέλος θα ήθελα να ασχοληθώ με το ζήτημα της ε, χώρας καταγωγής του πολιτιστικού αγαθού. Όταν αυτή δεν μπορεί να προσδιοριστεί, πιστεύουμε ότι όταν δεν προσδιορίζεται η χώρα καταγωγής, η χώρα προέλευσης, η άδεια θα πρέπει να συνοδεύεται με συνοδευτικά έγγραφα και αποδεκτικά στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι τα πολιτιστικά αγαθά εξήκτησαν από την χώρα εξαγωγή σύμφωνα με του δικού τη νόμου και κανονισμού. Ανεπομονούμε να κάνουμε τη συζήτηση με τους κοιόδους και σα ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σα. Ευχαριστούμε. Μιλήσατε για το Άλντε γενικότερα. Να δώσω λοιπόν το λόγο τώρα στον κύριο Σόλτσο, ο οποίο θέλει να μιλήσει εκ μέρου τη ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Θέλω να σε μιλήσω αντί για την κυρία Φορέντζα που είναι σκιώδη συζητήτρια. Και. Ακριβώς είπαμε κατά την παρουσίαση. Θεωρεί πάρα πολύ θετική την πρωτοβουλία της Κομισιόν όσον αφορά την εισαγωγή των πολιτικών αγαθών. Ευχαριστούμε τους ε, συνεισηγητές για το σχέδιο κειμένου. και εμείς ε, δηλώνουμε ότι θα συνεργαστούμε. Ίντερπολ λέει ότι η μαύρη αγορά για τα πολιτικά αγαθά είναι τόσο επικερδής όσο το λαθρεμπόριο όπλων ή ναρκωτικών. Και δυστυχώς ο βασικός προορισμός είναι η Αμερική, η ΙΠΑ και η Κίνα. Και υπήρχε συνένεση μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Και θα πρέπει αυτά τα 200 χρόνια προβλέπονται από την στιγμή της εισαγωγής να μειωθούν. Σύμφωνα με το άρθρο 5 έχουμε κάποια συγκεκριμένα αγαθά εδώ και θα πρέπει να δούμε αν αυτό είναι το πιο σωστό μέσο και αυτή η διπλή διαδικασία για την άδεια εισαγωγή θα πρέπει να δούμε πώς θα διατυπώσουμε καλύτερα αυτόν τον κανόνα. Εμείς θα συμβάλλουμε με κάποιες τροπολογίες και όπως είπαμε θα συνεργαστούμε για αυτό το σημαντικό θέμα. Τώρα, δεν είναι εδώ ο επόμενο ε, ομιλητή και ο Σβέντα και τώρα ο κύριο Μπούχνερ. Ευχαριστώ ε, πολύ και τους δύο εισηγητές. Ε, θα ήθελα αρχικά να τονίσω ότι η πρόθεση της ε, Κομισιόν ε, υποστηρίζεται, την υποστηρίζουμε απολύτως και αυτό σημαίνει ότι ε, δεν επικεντρωνόμαστε μονάχα στην χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αλλά γενικότερα στην καταπολέμηση παράνομων δραστηριοτήτων και φυσικά του ξεπλήματος. Τώρα όσον αφορά ε, τα πολιτιστικά αγαθά θα ήθελα να πω κάτι το οποίο υπόθηκε πολλές φορές. Το θέμα δεν αφορά μονάχα ε, της αρχαιότητας ε, και ένα όριο 250 χωρών, χρόνων αλλά υπάρχει και η σύγχρονη τέχνη υπάρχουν σύγχρονα δημιουργήματα τα οποία είναι πολιτιστικά αγαθά ε, και εδώ λοιπόν ε, θα ήταν παράλογο να έχουμε το όριο των 250 ε, χρόνων και εδώ λοιπόν μπορεί ε, να υπάρξει μεγάλη χειραγώγηση και απάτη. Είναι σημαντικό επίσης ε, η διαμετακίνηση να ρυθμιστεί, διότι εκεί υπάρχει πραγματικά η δυνατότητα να σταματήσουμε παράνομες ε, δράσεις και αυτό το έχουμε επιτύχει σε άλλους κανονισμούς όπως είναι για παράδειγμα στο κανονισμό για το dual use την σύμβαση της Μάλτας επίσης είναι ε, εφικτό και θα πρέπει να γίνει Ιδιαιτέρως ε, η αστυνομία στις χώρες προέλευσης είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός, όχι μονάχα τα τελωνία, διότι η αστυνομία γνωρίζει ε, τους δρόμους του παρόνιμου εμπορίου οι, άδειε εισαγωγών είναι πολύ σημαντικό ε, για εμάς. Ε, είναι κάτι τέτοιο είναι αναφίβολο. Ευχαριστώ πολύ και ε, ανυπομονούμε στη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Και για το EFTT η κυρία Μπεγκίν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Διάβασα με προσοχή την εκθέσή σας. Σας ευχαριστώ κύριε Σύγητες. Όπως έχω πει πολλές φορές αυτά τα πολιτιστικά αγαθά από τη Συρία και το Ιράκ δεν εμπίπτουν σε καμία ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έχει φτάσει λοιπόν η στιγμή να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ τους συνεισηγητές επειδή έλαβαν υπόψη και μια από τις δικές μου ανησυχίε την ομοιομορφία των τελωνιακών ελέγχων. Εγώ ασχολήθηκα πολλές φορές με αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για κοινή εμπορική πολιτική χωρίς τέτοια ομοιομορφία των ελέγχων και όσον αφορά τα πολιτιστικά αγαθά παρατηρείται port shopping. Για να λειτουργήσει ο κανονισμός ε, αυτός θα πρέπει να είναι ένας από τους κύριους τομείς που θα παρέμβουμε. Στον τελωνιακό τομέα είναι επίσης σημαντικό να ληφθεί υπόψη και άλλη μια σύσταση που θα βοηθήσει στην άρση της γραφειοκρατίας να υπάρξει ηλεκτρονικό μητρό. Δεύτερον, εκτιμώ ιδιαίτερα την τεχνική υποστήριξη που θα παρασχεθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να μπορέσει να τηρηθεί αυτός ο κανονισμός όταν θα τεθεί σε ισχύ. Ταυτόχρονα, θεωρώ ότι μπορεί να βελτιωθεί και άλλο αυτή η πρόταση. Όπως είχα προβλέψει στην πρώτη μας ανταλλαγή απόψεων, θέλω να έχουμε ένα σαφή ορισμό του πολιτιστικού αγαθού που να ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Επίσης, θα ήθελα να εμβαθύνουμε το ζήτημα της ηλικία των πολιτιστικών αγαθών και θα υποβάλω σχετικέ τροπολογίε. Η νόμιμη αγορά πολιτιστικών αγαθών δίνει δουλειά σε 350.000 ανθρώπους στην Ευρώπη και 90.000 ε, ε, παραπλεύρος ε, πρέπει να αποφύγουμε καταχρήσεις και οτιδήποτε άλλο μπορεί να επηρεάσει τη δουλειά αυτών των ανθρώπων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Βλέπω ο κύριος David Campbell έχει μόλις ε, φτάσει. Θα ήθελα να δώσω λοιπόν αμέσως το λόγο. Σας ευχαριστώ. Συγγνώμη. Είχε κίνηση, έχασα για ένα τρένο και ξανά είχε μετά κίνηση. Θα τα ξέρετε. Ήθελα ε, να σας πω ότι γενικώ καλά τα λέει αυτό το κείμενο, αλλά προσοχή να μην υπερβάλλουμε όσον αφορά τη γραφειοκρατία που είναι η προϋπόθεση της εφαρμογής. Και είναι θέμα αυτό το κατόφλι με τα χρόνια που πρέπει να περάσουν. Και το θέμα είναι πώς μπορεί να αποδείξει κανείς πόσο αρχαίο είναι ένα αντικείμενο. Να, που επισέρχεται η γραφειοκρατία. ερώτηση. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε πριν ανοίξουν τα σύνορα άρθρα 4-5, το ηλεκτρονικό σύστημα, όπως έχουν πει οι συνεισηγητές, είναι ένα σωστό βήμα και επίσης για τις μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουν τους πόρους να κάνουν αυτά που πρέπει. Άρα και εδώ είναι θετική η ρύθμιση. Δεν ξέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει να χρειάζονται πλέον πόροι όσον αφορά τις αρχές, τα τελωνία. Δημοσιονομικά ποιε θα οι επιπτώσει. Τι θα γίνει όταν μια χώρα προέλευση δεν μπορεί να εντοπιστεί και δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι τα εμπορεύματα, τα αντικείμενα αυτά τέλο πάντων να σχοληθούν νομίμω στην προηγούμενη χώρα. Η πρόεδρο, ε, νομίζω ακούσαμε όλου του χειρότερου συζητητέ. και ε, αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο που θέλει τον λόγο, που δεν νομίζω ότι ισχύει, τότε μπορούμε να τελειώσουμε με τις επεμβάσεις των ε, μέλλον Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ο κύριος Λάγκια. Μου απαντήθουν οι ερωτήσεις. Νικόλ από την ε, DG Taxud. Σε ευχαριστώ Πρόεδρε για το πρώτο θέμα, δηλαδή αν οι τολωνικές αρχές χρειάζονται περισσότερους πόρους για τους ελέγχους που προβλέπονται από το κείμενο ο στόχο δε όμως δεν είναι εκείνο. Είναι το πώς θα μπορούμε να έχουμε ελέγχου με τους πόρους που υπάρχουν σήμερα. Επίσης θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η πρόταση του κειμένου λέει ότι οι αρμόδιες αρχές θα αναλάβουν τους ελέγχους και θα πρέπει να έχουν τους αναγκαίου πόρους κλπ είναι ένα από τα στοιχεία που θα διευκολύνουν τους ελέγχους, δηλαδή αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα για να εφαρμοστεί το άρθρο 4 και το άρθρο 5. Εμείς μελετούμε το πώς θα βρεθεί κατάλληλη χρηματοδότηση για αυτό το σύστημα. Τώρα για το τι ισχύει όταν δεν ξέρουμε ποια είναι η χώρα προέλευση, δίνοντα κοιτάλια στην κυρία Μήτου, την συναδελφή. Ευχαριστώ. Όταν δεν μπορούμε επομένω να εντοπίσουμε τη χώρα προέλευση, το οποίο μπορεί να ισχύει για τα παλαιότερα πολιτιστικά αγαθά εδώ, υπάρχουν δύο εκδοχέ. Ή δεν γίνεται η εισαγωγή, Δεν θέλουμε να αποδειχθεί από πού ήρθε το, το προϊόν ή είμαστε ευέλικτοι. Και όταν η χώρα εξαγωγής, δηλαδή η τελευταία χώρα από όπου βγήκε το αγαθό και ήρθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν έχει προσυπογράψει την σύμβαση UNESCO του 70 γίνει χώρα, ε, τότε αυτό μπορεί να αρκέσει αν αυτός που έχει το αγαθό που ε, αποδείξει ότι νομίμως βρισκόταν εκεί το αντικείμενο. Είπαμε πάντως ότι στη χώρα εξαγωγής δεν θα πρέπει να είναι τα αγαθά μόνο για να επανεξαχθούν, δηλαδή να είναι μόνο τρανζιτή για για διαμετακόμιση. Θα πρέπει να έχουν μείνει τουλάχιστον τα επίμαχα αγαθά, τουλάχιστον ένα μήνα, να έχουν μείνει τόσο κάποιο χρονικό διάστημα την άλλη μεριά. Όντως ο, ο ένας μήνας παραμονής δεν αρκεί. Οπότε μελετούμε τη δυνατότητα να αυξηθεί ε, ο χρόνος παραμονής σε κάποια άλλη χώρα για πολύ περισσότερο διάστημα, Φερρυπίν για 10 χρόνια, Λάγκη. Σε, σε ευχαριστούμε πολύ. Άλλες ερωτήσεις προς την Επιτροπή. Όχι, επομένως, να ξαναδώσουμε το λόγο στους συνεισηγητές, ίσως αντιστρέφοντας την σειρά γιατί δίνοντας πρώτο το λόγο στον κύριο Ντάλτον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για απαντήσεις της Κομισιόν. Αποδεικνύουν πόσο δύσκολο είναι τα θέματα που μας απασχολούν. Να είμαστε προσεκτικοί για την ηλικία, για την αξία, τα κατόφλια αυτά. Να, Εάν η ηλικιακή απέτηση κατέβει τότε μπορεί να έχουμε ένα βιβλίο που το γράψει ας πούμε για τον πρώτο παγκόσμιο παππούς μου το παίρνω στις διακοπές μου στις ήπα ε, και μετά το αφήνω το ξαναφέρω στο σπίτι ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τι θα γίνει με αυτό. Επίσης τι θα κάνουν τα τελωνία. Πώς θα βρουν την αξία την ηλικία. Άρα να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πώς θα ρυθμιστούν όλα αυτά. Βέβαια, αν κανείς καταλάβει ποιο είναι το θέμα, ποιο είναι το ζουμί, τότε βρίσκει και τους κανόνες. Εδώ θα βάλω τελεία, αλλά βέβαια έχουμε σύντομα την ε, προθεσμία για τις τροπολόγιες. Και δεν είναι θέμα ότι διαφόρησα εγώ με τη σύνηση γήτρια. Η κάθε ομάδα έχει τις δικές της απόψεις. Κάθε πολιτική ομάδα. Ναι, Εμεί τέλο πάντων θέλουμε να συγκεράσουμε όσο γίνεται περισσότερε απόψει. Και πιστεύω και η κυρία Μόσκα το ίδιο πρέσβευε. Οπότε με όλες αυτές τις τροπολογίες θα δουλέψουμε. Αλέσια Μόσκα έχεις το λόγο. Ευχαριστώ και εγώ συμφωνώ με το στόχο που ανέφερε ο συνεισηγητής μου. Θέλω να ξεκινήσω από τα κοινά στοιχεία που προκύπτουν από τη συζήτηση που κάναμε. Πρώτα απ' όλα είναι σαφές ότι ε, με το στόχο συμφωνούν όλες οι πολιτικές ομάδες. Να υπάρχει δηλαδή ένας κανονισμός ο οποίος θα μας δώσει τη δυνατότητα να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά το παράνομο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών. Επίσης ε, συμφωνούν όλοι ότι ο κανονισμός αυτός ε, δεν θα πρέπει να επιβαρύνει υπερβολικά τους φορείς του τομέα. Μεταξύ όλων των απόψεων λοιπόν που ακούσαμε στη σημερινή συζήτηση και που έχουμε συναντήσει στη συζήτηση των τελευταίων εβδομάδων θα πρέπει να βρούμε ποιες ε, λύσεις ε, υπάρχουν που τεχνικά να μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αναφέραμε. Ουσιαστικά πρέπει να δούμε και τα πιο ακαθόδη ζητήματα, την ηλικία, το κατόφλιο ηλικίας, ε, τη χώρα προέλευσης και πώς θα καταρτήσουμε τον κατάλογο των αγαθών αποτελεσματικά. Ε, βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών. Ένα από αυτά τα στοιχεία και ένα από τα πιο επίμαχο προκύπτει ότι είναι το θέμα του κατοφλίου ηλικία, το όριο ηλικία, όπω είδαμε. Και για να απαντήσω στον συνεισηγητή και στην ένστασή του, αν πάμε να μειώσουμε ναι, αυτή την ηλικία θα αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα, αλλά το να προσθέσουμε την αξία του αγαθού που κινείται εμπορικά θα βοη... λειτουργήσει ως εγγύηση. Διότι όταν εμείς έχουμε ε, ε κάποιο αντικείμενο πολύ ψηλή αξίας πάνω μας, αυτό συνοδεύεται εξορισμού με διάφορα έγγραφα, περισσότερο που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Πιστοποιήσεις, ε, Οπότε δεν θα επιβαρύνει αυτό ιδιαίτερα τους φορείς. Από μόνο τους τα αγαθά αυτά συνοδεύουν ήδη ένα τέτοιο αγαθά το οποίο κυκλοφορεί νόμιμα. Οπότε θεωρούμε ότι εδώ έχουμε ένα παράδειγμα του πώς θα μπορούσαν να βρεθούν ε, λύσεις οι οποίες θα ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσει. Εγώ έχω σημειώσει, έχουμε σημειώσει όλες τις παρατηρήσεις που έγιναν και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να βρούμε μια λύση για όλα τα τεχνικά προβλήματα που έχουν προκύψει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τους ε, δύο εισηγητές. Καλό θα ήταν φυσικά στο Κοινοβούλιο να επιτύχουμε πλειοψηφία για την έκθεση. Αυτό θα ενισχύσει τη δική μας θέση ε, και στο Συμβούλιο. Κύριε θέλετε να κλείσετε. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Συμπρόεδρε. θέλετε να κλείσετε τη συνεδρίαση. Ναι, ευχαριστώ. Πολύ ευγενικό εκ μέρου σα. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών σε δύο μέρε 25 Απριλίου το μεσημέρι. 12 ώρα το μεσημέρι. Δεν απομένει πολύς χρόνος λοιπόν. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσουμε αυτή την κοινή συνεδρίαση και να ευχαριστήσω τον συμπροεδρό μου τον κύριο Λάγκη, και θα επανέλθουμε για την εξέταση των τροπολογιών των Ιούνιων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Συμπρόεδρε. Εδώ ολοκληρώνεται το σημείο 7 και το επόμενο σημείο είναι η συνάντηση των συντονιστών που θα πραγματοποιηθεί και κλεισμένων των θυρών και θα ξεκινήσει σε 10 λεπτά.